Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να καλωσορίσω στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπή μα. Ο πρόεδρος κύριος δεν ε, μπορεί Δυστυχώ να είναι παρόν στην ε, δική μα συνεδρίαση λόγω λιμένων υποχρεώσεων. Κατόπιν τούτου έχω την ε, χαρά να τον ε, αναπληρώνω και να προεδρεύω σε αυτή τη συνεδρίαση της επιτροπή Ελέγχου Προεπολογισμών. Ευθύ εξ αρχής θα ήθελα να πω το εξή. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης είναι η έγκριση αυτής στις 11 Μαΐου λάβατε το σχέδιο της σημερινής διάταξης και αν δεν έχετε παρατηρήσεις, ε, θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Κατόπιν νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο σημείο που είναι οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου. ερμηνεία έχουμε σε 16 γλώσσες που σημαίνει ότι οι συνάδελφοι μπορούν ε, να ακούσουν και να μιλήσουν 16 γλώσσες. Και θέλω επίσης να σας ε, επισημάνω ότι η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Κατά τα άλλα, ε, για σήμερα προβλέπονται επίσης ηλεκτρονικές ε, ψηφοφορίες που σημαίνουν σας παρακαλώ πολύ να έχετε ε, μαζί σας την ηλεκτρονική σας κάρτα για τις ψηφοφορίες. Αύριο στις 25 Μαΐου προβλέπεται άλλη μία συνάντηση με τους εκπροσώπους του ελεγκτικού συνεδρίου. Και στη συνάντηση αυτή θα λάβει μέρος και ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου, ο κύριο Μπούζεκ. Στη συνεδρίαση αυτή ε, θα προεδρεύσει ο αντιπρόεδρο μα κύριο jean Οντί. Πάλι αύριο, για αύριο, στην αυριανή ημέρα αναφέρομαι. Στις 6 ώρα θα έχουμε μία μικρή δεξίωση στο κτίριο PHS ε, με όσους θα συμμετάσχουν αύριο στην κοινή αυτή συνεδρίαση. Μετά λοιπόν τις ανακοινώσεις του Προέδρου νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στην έγκριση των πρακτικών της 28ης Φεβρουαρίου, της 22ης Μαρτίου και της 28ης Μαρτίου 2011. Ε, Αν δεν έχετε παρατηρήσεις για τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων μέχρι το τέλος της ημέρας, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται τα πρακτικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα λοιπόν ας περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι ο διορισμός μέλους ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι Σουηδικές ε, αρχές ε, πρότειναν τον κύριο Hans Gustav Westberg Η διαδικασία προβλέπει ότι ε, πριν από ε, τον διορισμό του υποψηφίου για το ελεγκτικό συνέδριο θα προηγηθεί ακρόαση. Κατά τα άλλα, στο ενημερωτικό δελτίο Κοκομπού, στο Info, εκεί υπάρχει ε, ένα λάθος. Αναφέρεται ότι η τελική ψηφορία θα γίνει στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Προφανώς αυτό είναι λάθος εκ παραδρομής και η τελική ψηφορία θα γίνει στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Μετά από αυτήν την ακρόαση ε, και κλεισμένων των θυρών θα αποφασίσουμε, θα τοποθετηθούμε για αυτόν τον υποψήφιο και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο στον υποψήφιο τον κύριο Hans Gustav Westberg ο οποίος θα απαντήσει στις ε, ερωτήσεις ε, που του υποβάλαμε και θα τοποθετηθεί και αυτός θα εκφράσει την άποψή του αυτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε και προτού σας ξαναπώ ολόκληρο το βιογραφικό μου, σας πω μερικά πράγματα για τον εαυτό μου. Είμαι 59 ετών. Αυτό σημαίνει ότι έχω επαγγελματική καριέρα λίγο πάνω των 30 ετών. Και έχω ένα μεικτό ε, μια μεικτή σταδιοδρομία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Η μισή μου καριέρα ήταν στο δημόσιο τομέα και η υπόλοιπη μισή στον ιδιωτικό. Τουλάχιστον στη δικιά μου χώρα αυτό είναι σχετικά σύνηθες, δηλαδή το να πηγαίνει κανείς από τον ένα τομέα στον άλλον, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια προστιθαμένη αξία στην όλη μου εμπειρία. Επίσης υπήρξα δραστήριο στην πολιτική για περίπου 15 χρόνια ε, ήμουν εκτός πολιτικής όταν ήμουν δημόσιος υπάλληλος, διότι δεν θεωρώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι ενεργοί στην πολιτική όσο υπηρετούν στο δημόσιο. Αυτή τώρα η μετακίνηση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα πιστεύω ότι με βοήθησε να αποκτήσω αξιόλογη εμπειρία. Δηλαδή, αν θέλετε, υποφελήθηκα πολύ από την μεταβολή του προσανατολισμού της σταδιοδρομίας μου. Ε, υπάρχουν και ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Ε, αλλά και για τους και τους δύο τομείς υπάρχουν ορισμένες βασικές αξίες καλής διοίκησης. Και θα μπορούσα να πω ότι αυτές οι αξίες είναι η εξοικονόμηση, η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία, η διαφάνεια, το ανοιχτό μυαλό και βεβαίως οι στόχοι που είναι σωστά προσδιορισμένοι ε, και επιδιωκόμενοι. Στον δημόσιο τομέα τις περισσότερες φορές ε, η διαφάνεια είναι καλύτερη από στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ στον ιδιωτικό τομέα συνήθως οι στόχοι είναι καλύτερα προσδιορισμένοι. Όπως μπορείτε να δείτε λοιπόν από το βιογραφικό μου, έχω μακρά εμπειρία στα διοικητικά. Ήμουνα ε, γενικός διευθυντής και αναπληρωτής σε κυβερνητικό φορέα και πρόσφατα υπήρξα και υφυπουργό σε διάφορα υπουργεία. Το πιο σημαντικό ήταν ότι ήμουν παρά το Πρωθυπουργό. Σε όλες αυτές λοιπόν τις ε, θέσεις, τις υψηλές θέσεις διοίκησης, είχα τη δυνατότητα να εφαρμόσω αυτές τις αξίες. Ακόμη όμως έμαθα και τη σπουδαιότητα του ελέγχου και του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ακόμη είμαι πεπισμένος για τη σπουδαιότητα του ευρωπαϊκού σχεδίου και το σημαντικό ρόλο που το ελεγκτικό συνέδριο παίζει για να έχει αξιοπιστία η Ένωση προς τους πολίτες. Λοιπόν, αν διοριστώ μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, νομίζω ότι θα μπορέσω να προσφέρω το κριτικό οφθαλμό, αν μπορώ να το πω αυτό, από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τη μακρά μου εμπειρία. Ελπίζω ότι με αυτή την εμπειρία μου θα μπορέσω να συμβάλλω στο έργο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο έχει πολλά σπουδαία πράγματα να κάνει. Οπωσδήποτε χρειάζονται πολιτικοί στόχοι σαφείς και υλοποιήσιμοι. Ακόμη είναι απαραίτητο να υπάρχει σωστή λογοδοσία για την δαπάνη των κονδυλίων των ευρωπαϊκών πάλι. Είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των δαπανών ώστε να προστατεύσουμε τα χρήματα των φρολογούμενων. Ακόμη πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να έχει και έχει μία στρατηγική για να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα από τους ελέγχους και για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας σωστά τους πόρους. Αυτό το έργο του συνεδρίου είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ε, Κοινοβουλίου, Εθνικών Κυβερνήσεων, και εθνικών ελεκτικών αρχών. Είμαι στη διάθεσή σας τώρα για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βέσπερκ, ε, είσαστε ενδιαφέρον υποψήφιος ε, για το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί πράγματι εσείς έχετε περάσει και από τους δύο τομείς, και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα και έχετε εντυπωσιακό βιογραφικό. Στο τέλος ήσασταν στο κέντρο πολιτικής εξουσίας ε, της Σουηδίας. Εγώ δεν διαβάζω σουηδικές εφημερίδες όπως το κάνει στην αδελφό μου από την Ισπανία και δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε εκεί, όμως θεωρώ ότι έχετε πλούσια εμπειρία. Είσαστε πολύ ενδιαφέρον υποψήφιος και αυτό το είπα ήδη. Εσείς ο ίδιος επισημάνατε το ότι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των ε, δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κέριο σημείο. Και γι' αυτό σας ερωτώ, ως κάποιος ο οποίος γνωρίζει τον ιδιωτικό τομέα και κατόπιν τούτου γνωρίζει και το θέμα της αποτελεσματικότητας, αλλά παράλληλα είναι εξοικειωμένο και με την πολιτική, κατά την άποψή σας, πού ακριβώς εντάσσεται ο ρόλος του ελεγκτικού συνεδρίου, κυρίως όταν πρόκειται για την αξιολόγηση αξιολόγηση της απόδοσης, δηλαδή σωστή χρήση και αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με άλλα λόγια, ευρωπαϊκή υπεραξία. Σύντομα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια έκθεση αξιολόγησης. Κατά την άποψή το ελεγκτικό συνέδριο τι ρόλο μπορεί να παίξει σε όλο αυτό το πλαίσιο. Πολύ ωραία. Ο κύριος Φιέρνα. Πρόεδρε. Κύριε Βέσπερκ, νόμιζω ότι το βιογραφικό σας είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αλλά σαν πρώην επικεφαλής των λογιστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με σταδιοδρομία ε, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, νομίζω ότι δεν έχετε γνώσεις λογιστικές σύμφωνα με το βιογραφικό σας. Σε σχέση λοιπόν με αυτό το ζήτημα αναρωτιέμαι αν έχετε διαβάσει την πρόσφατη έκθεση του ελεκτρικού συνεδρίου, την Draft Assurance Report. Ποια είναι, ε, αν το έχετε διαβάσει, τι νομίζετε, ε, είναι θετική ή αρνητική η γνώμη τους, διότι για μας το Ευρωκοινοβούλιο ε, το να δώσουμε απαλλαγή για να δώσουμε μάλλον απαλλαγή, είναι πολύ σημαντικό να βασιστούμε στη γνωμοδότηση του λεγκτικού συνεδρίου. Και είναι πολύ σημαντικό οποιοδήποτε νέο μέλος να αντιλαμβάνεται τους στόχους του Draft Insurance Report, αυτής της έκθεσης. Έκθεση αξιοπιστίας, ενδεχομένως. Κύριε Βέσπερκ, ε, η δική μου ερώτηση είναι παραλλαγή της ερώτησης κυρίας Αντρέσεν. Δηλαδή, εγώ δεν ανησυχώ τόσο πολύ στην περίπτωση κατά την οποία το ελεγκτικό συνέδριο έχει μέλη ...στον οποίο το βιογραφικό δεν αναφέρεται ότι είναι εξέχοντες και επαΐοντες ε, λογιστές είναι δυνατόν και γιατί όχι το ελεγκτικό συνέδριο να έχει μέλη που να προέρχονται από διαφορετικούς και άλλους τομείς ε, γνώσεων. Όμως ε, όσον αφορά τους ε, τελευταίους υποψήφιους που είδαμε σε αυτές τις τελευταίες μας θητείες οι περισσότεροι πρέπει να πω είχαν σαφείς γνώσεις δημόσιων λογιστικών. Και γι' αυτό λοιπόν ερωτώ εσάς το Ευρωπαϊκό Συνέδριο πρέπει να επιμένει στο να υπάρχουν ειδικέ γνώσεις λογιστικής ή όχι. Και κατά την άποψή σας πόσα από τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου θα έπρεπε να μπορούν να, έπρεπε να επιδεικνύουν αυτές τις ειδικέ γνώσεις. Πολύ ωραία. Ε, κύριε Βαϊσπέρκα, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την ερώτησή σας για την απαλλαγή μου όταν ήμουν διευθύνων σύμβουλος. Ε, πρόκειται για μια εξωτερική ελεγκτική εταιρεία που υπέβαλε έκθεση στην ετήσια συνεδρίαση, τη Γενική Συνέλευση δηλαδή, του αντίστοιχου ΣΕΒΑ της Σουηδίας και μου δόθηκε απαλλαγή και τις δύο φορές. Ήμουν διευθύνων σύμβουλος αναπληρωτή στον πρώτο χρόνο και στη συνέχεια στο τέλος της ε, ζωής αυτού της οργάνωσης ήμουνα τέσσερις μήνες διευθύνων σύμβουλος και μου δόθηκε απολογή και στις δύο περιπτώσεις. Στη συνέχεια συγχωνεύτηκε με άλλον οργανισμό. Τώρα, όσον αφορά το έργο μου στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τις απόψεις μου σε σχέση με τις εθνικές τοποθετήσεις. Όπως ξέρετε, η Σουηδία έχει τοποθετηθεί θετικά όσον αφορά τις εθνικές δηλώσεις της και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό. Ε, είναι ανοιχτή ε, και η δήλωση αξιοπιστίας ήταν πολύ θετική. Όσον αφορά τώρα την διαχείριση της κρίσης, δεν ήμουν υπεύθυνο αυτού του οργανισμού όταν εμφανίστηκε το τσουνάμι, αλλά η αξιολόγηση μετά την κρίση κατέδειξε ότι η σουηδική κυβέρνηση και το γραφείο του Πρωθυπουργού χρειαζόντουσαν ένα φορέα οργανισμού της κρίσης που δεν υπήρχε. Αυτό ήταν το συμπέρασμα δηλαδή από την διαχείριση της κρίσης. Το συμπέρασμα μας βασικά ήταν ότι δεν αντιδράσαμε αρκετά γρήγορα όταν μας χτύπησε η κρίση χωρίς να το αναμένουμε. Το γεγονός ότι υπήρχαν χιλιάδες Σουηδοί τουρίστες στη νότιο-ανατολική Ασία μας διέφυγε όταν σχεδιάσαμε το σύστημα διαχείρισης κρίσεων. Γι' αυτό ακριβώς αποφάσισε η ε, κυβέρνηση να δημιουργήσει έναν νέο οργανισμό και σαν υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό ήταν δικά μου δουλειά να οργανώσω αυτό τον οργανισμό. Η απόφαση ήταν δικιά μου, ήταν της κυβέρνησης, αλλά η οργάνωση του φορέα ήταν δικιά μου ευθύνη. Οργανώσαμε λοιπόν ένα φορέα που παρακολουθεί συνεχώς 365 μέρες το έτος όλο το 24ωρο την εξέλιξη των προγραμμάτων και επίσης αναπτύξαμε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και δημιουργήσαμε ακόμη τη δυνατότητα για αυτόν τον φορέα να είναι όχι whistleblower δεν είναι σωστή λέξη ε, δεν καρφώνει αλλά επαγρυπνεί και προειδοποιεί. Το σφυδικό σύστημα είναι σχετικά αποκεντρωμένο και οι φορείς έχουν δικιά τους ευθύνη να ενεργήσουν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ήταν απαραίτητο να δημιουργήσουμε αυτόν τον φορέα που παρακολουθεί τα πάντα επί 24 ώρου βάσης και προειδοποιεί. Ακόμη δώσαμε τη δυνατότητα σε αυτό τον φορέα να λαμβάνει κάποιες αποφάσεις σε περίπτωση που η κρίση εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα χρηματικό αν θέλετε διότι το πρόβλημά μας με το τσουνάμι δεν ήταν ότι είχαμε έλλειψη χρημάτων, είχαμε όλους τους πόρους διαθέσιμους. Απλώς δεν χρησιμοποιήσαμε τους πόρους όπως ήταν απαραίτητο. Ε, και γι' αυτό χρειάστηκε να δημιουργεί νέος φορέος υπεύθυνο για την απόκριση στην κρίση. Έχουμε δοκιμάσει λοιπόν τις δυνατότητες αυτού του φορέα σε κρίσεις όχι τόσο μεγαλός αυτή με το τσουνάμι, αλλά όταν είχαμε την γρήπη των χείρων, στην Ευρώπη πριν από ένα χρόνο παν, ε, δοκιμάστηκε η λειτουργία αυτού του φορέα καθώς και ε, σε μικρότερες περιπτώσεις όπως καταιγίδων ή εθνικών καταστροφών άλλων τύπων και πρέπει να πω ότι λειτουργεί σχετικά καλά. Και είμαι πολύ περήφανος να σας πω την αλήθεια για τη σύσταση αυτού του φορέα. Ακόμη, με ρωτήσατε για κάποιους ισχυρισμούς για πάτη ε, κατά τις εκλογές. Θα ήθελα να επεκταθώ λίγο πάνω σε αυτό το θέμα γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο να έχει κανείς όλα τα δεδομένα όταν διαβάζει μόνο μία ή κάποια εφημερίδα από τη Σουηδία. Οι ισχυρισμοί λοιπόν ήταν ότι στις... πριν από τις εκλογές στο περιφερειακό επίπεδο στη Σουηδία δηλαδή σε εκλογές Landsdienen όπως τις αποκαλούμε. Λοιπόν, οι ισχυρισμοί ήταν ότι σε αυτό το επίπεδο είχα επιτρέψει εξαπάτηση στην ε, μέτρηση των ψήφων της προκαταρτικής ψηφοφορίας στο κόμμα μου. Αυτός ήταν ο ισχυρισμός για το 2001. Όμως το 2001 δεν έγινε καμία τέτοια προκαταρκτική ψηφοφορία. Το 2002 έγινε αυτή η προκαταρκτική ψηφοφορία. Κάποιος δεν κατάλαβε κάτι λοιπόν πολύ καλά. Δεύτερον, εγώ ο ίδιος δεν ήμουν υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Ουσιαστικά δεν είχα υπάρξει υποψήφιος σε εκλογές για 10 χρόνια. Λοιπόν, δεν είχα τίποτα να κερδίσω απέρριψα αυτούς τους ασχερισμούς. Ε, είπα και ξαναλέω ότι δεν γνωρίζω να έχει υπάρξει οποιαδήποτε εξαπάτηση κατά τις ε, προκαταρτικές μας εκλογές. Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε τέτοιες δραστηριότητες και δεν έχω επιτρέψει ποτέ τέτοιες δραστηριότητες. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το ρόλο του ελεκτικού συνεδρίου όσον αφορά την, ε, τον έλεγχο της αποδοτικότητας. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι δεν είμαι ακόμη μέλος ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά η εμπειρία μου από τον ιδιωτικό τομέα και από το δημόσιο τομέα μου λέει το εξής. Βεβαίως ο έλεγχος που έχει σχέση με την απαλλαγή είναι πάρα πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα για το κοινοβούλιο. Χρειάζεστε πολύ σημαντικές πληροφορίες για να μπορέσετε να δώσετε την απαλλαγή. Νομίζω όμως ότι ο έλεγχος της αποδοτικότητας και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Αν πραγματικά θέλετε τα χρήματά σας να αποδώσουν, αν θέλετε να προστατεύσετε τα χρήματα του φορολογούμενου, αν θέλετε να προσθέσετε ε, να έχετε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην χρήση των κοντιλίων. Κατά την άποψή μου λοιπόν ο έλεγχος της αποδοτικότητας αυξάνει σε σπουδαιότητα και θα ήταν πολύ χρήσιμο να μετακινηθούν κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχω διαβάσει πολλά πράγματα από το ελεγκτικό συνέδριο, το ευρωπαϊκό ακόμη. Οι ειδικέ εκθέσεις που έχω διαβάσει πάντως είναι πολύ συγκεκριμένες και νομίζω ότι ακριβώς αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο. Να είναι συγκεκριμένες οι τοποθετήσεις. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τη σπουδαιότητα της απαλλαγής. Αυτά, κάτι τέτοιο θα ήταν προβληματικό. Για να λύσουμε το πρόβλημα βεβαίω πρέπει να ενισχύσουμε την αποδοτικότητα στο ελεκτικό συνέδριο. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική παράμετρος και θα ήταν σημαντικό μέρος της εργασίας μου σαν μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ε, αν γίνω. Τώρα θα μιλήσω σβηδικά. Με ρωτήσατε λοιπόν γιατί ήθελα να γίνω μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, γιατί ζήτησα να είμαι υποψήφιος. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε επί μακρόν, Κριστόφ. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής. Για πολλά χρόνια είχα την άποψη ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο ήταν το πιο σημαντικό σχέδιο των τελευταίων ετών. Άλλωστε, προσπάθησα να παροτρύνω τη Σουηδία για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πιο σημαντική απόφαση που ελήφθη στη Σουηδία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ευρωπαϊκό σχέδιο όμως αυτή τη στιγμή εμφανίζει ανεπάρκειες και κενά. Πρώτα απ' όλα έχουμε έλλειψη αξιοπιστίας των πολιτών προς τους ηγέτες. Δεν έχουν επίσης εμπιστοσύνη στα χρηματοοικονομικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, είναι πεπισμένοι οι πολίτες για τη βέλτιστη χρήση αυτών των κοντιλίων Συνεπώς, ε, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. Αν γίνω λοιπόν, όπως ελπίζω, μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, θα χρησιμοποιήσω την πείρα μου των 30 ετών για να μπορέσω να συμβάλλω ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, να ενισχύσω την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τώρα, ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Ε, σε προηγούμενη ερώτηση είπα ότι ο έλεγχος των κονδυλίων είναι βεβαίως πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερα μέσα για αυτόν τον έλεγχο. Όλοι οι οργανισμοί μόνιμα πρέπει να βελτιώνουν την εσωτερική τους αποδεκτικότητα και την δράση τους. Δεν αποτελεί εξαίρεση το ενεγκτικό συνέδριο της Ευρώπης. Πρέπει να αναδιπλώσει τις, ε, τους διοικητικούς του πόρους, να τους ανακατανείμει μάλλον, ώστε να μπορέσει να ενισχύσει τις έρευνες και τους ελέγχους. Άλλωστε νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει. Οι έρευνες έχουν πολύ συμβάλει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του ελεκτικού συνεδρίου, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτό θα το δούμε μελλοντικά. Όσον αφορά τώρα την αντάσ, την ντάς, δηλαδή την δήλωση αξιοπιστία, ουσιαστικά είναι μια απαλλαγή αυτή. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά το έργο της, του ελεγκτικού συνεδρίου. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για μας είναι πολύ σημαντική. Αυτό αιτιολόγησε την τοποθέτησή μας. Και ξαναπαρνάω τώρα στα αγγλικά. Βεβαίω, ποτέ δεν υπήρξα ελεγκτή όπω είπατε. Είναι προφανέ αυτό από την, το βιογραφικό μου. Αυτό το οποίο φέρνω είναι μια μακρά διοικητική διευθυντική εμπειρία. Βεβαίως, στη διάρκεια αυτών των 30 ετών έχω συνεργαστεί συνεχώς με ελεγκτές και ε, λογιστικούς ειδικού στα λογιστικά. Η αποτελεσματικότητα και η εξοικονόμηση μπορούν να συμβάλλουν πολύ και αυτές τις εμπειρίες τις έχω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί ειδικοί στα λογιστικά μέσα στο πλαίσιο του ελεγκτικού συνεδρίου και μπορώ θαυμάσια να συνεργαστώ μαζί τους. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είμαι εγώ ειδικό. Επίσης, μια... με ρωτήσατε πόση εμπειρία πρέπει να έχει κανείς με τη λογιστική για το ελεγκτικό συνέδριο. Θα έλεγα ότι είναι σημαντικό πολλά μέλη να έχουν εμπειρία σε αυτό το τομέα, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει όλα τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου να προέρχονται από την λογιστική. Ευχαριστώ κύριε Βέσπεργα. Κοιτάξτε, οποτεδήποτε έχουμε εδώ μέλη του ε, υποψήφιους για το ελεγκτικό συνέδριο, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί θεωρούμε ότι ακόμα και αυτοί που δεν έχουν ειδικέ γνώσεις λογιστικής μπορούν να συμβάλλουν τα μάλα. Η Σουηδία είναι καθαρός συνεισφορέας ως χώρα και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί βεβαίως ε, πρέπει να ε, είμαστε υπόλογοι απέναντι στους πολίτες μας. Αυτό ισχύει και για τη Γερμανία. Θα τα έβρισκα ώρα πάρα πολύ καλά αν δεν είχατε πει, αν δεν είχατε πει ότι τις ειδικέ εκθέσεις τις βρίσκετε σωστές. Εγώ όμως δεν τις βρίσκω. Αυτές οι ειδικέ εκθέσεις για μένα δεν είναι σωστές και δεν βοηθούν σε τίποτα. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική που πρέπει να περιγράφεται στις ειδικέ αυτές εκθέσεις. Οι ειδικέ εκθέσεις ε, να προσφέρουν κάποιες λύσεις έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Κύριε Γιάλα